πολύ κυρίες και κύριοι. Τώρα περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου. Πρώτα απ' όλα, για... ο κύριος Καλινόφσκι για τα επενδυτικά ταμεία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα εναλλακτικά επενδυτικά ταμεία είναι πολύ σημαντικά για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και οι ε, διαχειριστές τους πρέπει να σέβονται τους κανονισμούς που επιτρέπουν να λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εποπτεία πρέπει να είναι αποτελεσματική για να μπορέσουμε να το επιτύχουμε αυτό. Θα πρέπει να καλύψουμε τα κενά στο ρυθμιστικό μας σύστημα και στο νομοθετικό μας σύστημα. Οι προτάσεις ε, οι οποίες ε, έχουν υποβληθεί βελτιώνουν τον τομέα και θα οδηγήσουν οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αξιοπιστία των θεσμών και γι' αυτό και όλες τις οικονομίες μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πυρίλο. Ο κύριο Πυρίλο έχει το λόγο. Ε, ε. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πυρίλο, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή ψηφοφορία δεν ένα σημαντικό βήμα μπροστά για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη ρύθμιση των ε, οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. Χάρη στην οδηγία, οι διαχειριστές αυτών των ταμείων θα πρέπει να καταγράφονται και να εξοδοτούνται και να σέβονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυστηρούς κανόνες ελέγχου. Όντω, είναι πρώτη φορά που το τομέα αυτό ρυθμίζεται και θεωρώ πω το έγγραφο που ψηφίστηκε θέτει του όρου για να φτάσουμε, ελπίζω, σύντομα σε μια πραγματική μια αγορά των ε, χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επέμεινε ώστε να υπάρξουν ισχυροί κανόνες για μεγαλύτερη εποπτεία της ε, χρηματοπιστωτικής βιομηχανίας που έτσι γίνεται και πιο ηθική. Το πρόσφατο παρελθόν της οικονομικής κρίσης που προκλήθηκε λόγω κερδοσκοπίας των, ε, των επενδυτικών ταμείων θα πρέπει να μας ε, βοηθήσει να στηρίξουμε αυτή την οδηγία για τη μεγαλύτερη προφύλαξη και προστασία των πολιτών. Εγώ υπερψήφισα και ζήτησα το λόγο για να συγχαρώ τον εισηγητή για τη δουλειά του. Ευχαριστούμε κύριε Πυρίλο. Ο κύριος Καμάλ έχει το λόγο τώρα. Κύριε Καμάλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όταν κοιτάξαμε την πρώτη αρχική πρόταση πριν 18 μήνες όλοι είχαμε απογοητευτεί διότι δεν μας είχαν συμβουλευτεί και θα ήταν ε, πολύ δύσκολη κατάσταση, θα είχε καταστρέψει τις αγορές και δεν θα μπορούσε κανείς ε, να επενδύσει σε μη ευρωπαϊκά ε, επενδυτικά θέματα ενώ χάρη στην εξαιρετική εργασία του Ευρωπαίου ε, του Επιτρόπου της Βελγικής Προεδρίας και των σκιωδών εισηγητών μπορέσαμε να βελτιώσουμε την κατάσταση για να μπορούν οι επενδυτές να συνεχίσουν να επενδύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με την ΕΣΜΑ ε, μπορέσαμε να έχουμε ένα συμβιβασμό που να ικανοποιήσει τους πάντες. Ευχαριστώ. Τώρα περνάμε στην ε, έκθεση του κυρίου μέρα και το λόγο έχει η κυρία Αντρικένε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, ε, για αυτό το πολύ ενδιαφέρον έγγραφο το οποίο είναι πολύ σημαντικό και τώρα η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια της ε, ε, καταργήσεως στην Ευρωπαϊκή Ενώσεως των ε, εμποδίων για την ελεύθερη διακίνηση στο στο χώρο Σέγγεν αντιλαμβανόμαστε ότι τώρα όλοι θα μπορούν να έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς βίζες χωρίς θεωρήσεις και κάτοικοι ε, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Κύπρου θα μπορούν να πηγαίνουν στην Ταϊβάν χωρίς θεώρηση και είναι μια εξαιρετική εξέλιξη στην οποία ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Λούνατσεκ και εγώ ε, εν ονόματι της πολιτικής μου ομάδος χαιρετίζω την κίνηση της Ταϊβάν για την ελεύθερη ε, άφηξη των ταξιδιωτών αλλά ε, νομίζω ότι ε, υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν αναγνωρίσει την Ταϊβάν ε, τι θα γίνει όμως με το κοσυφοπέδιο διότι 22 κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έχουν αναγνωρίσει το κοσυφοπέδιο και δεν έχει καν ξεκινήσει η συζήτηση με τη χώρα αυτή. Ελπίζω ότι η Επίτροπος Μάλστρομ επιτέλους θα κινητοποιηθεί για να μπορέσουν οι ε, κάτοικοι της χώρας αυτής να κινούνται εξίσου ελεύθερα με τους κατοίκους της Ευρώπης προς την Ταϊβάν. Τώρα το λόγο έχει σχετικά με την έκθεση Βαν Μπρέμ, την κυρία Εκ, για ένα λεπτό. Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω σου ειδικά. Το πρόγραμμα ανάκτησης το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάκτησης Ενέργειας ε, έχει στόχο να αυξήσει την επάρκεια σε ενέργεια και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα προγράμματα μπορούν να ξεκινήσουν πολύ γρήγορα και είναι πολύτιμα. Αυτή η συμφωνία Ε, επίσης υποχρεώνει σε χρήση της ε, σουηδικής αυτό είναι πολύ καλό βήμα. Θα μειωθεί η εξάρτησή μα από τις ε, τρίτες χώρες και με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να δουλεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρήματα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα τομέα να μετακινηθούν σε έναν άλλο τομέα, δηλαδή η αρχή των κυλιόμενων ε, κονδυλίων. Ε, το Συμβούλιο βέβαια ε, καθυστέρησε να το καταλάβει αυτό γιατί κάποια μεγάλα κράτη-μέλη έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μην τηρήσουν τις προηγούμενες τους υποσχέσεις αλλά είναι πολύ καλό που εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμείναμε και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων είπαμε ότι ήταν πολύ σημαντική η διαφάνεια και η απλοποίηση των ε, κανόνων και είμαι ικανοποιημένη που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέστησε σαφές ε, ότι θέλουμε να μειωθούν τα διοικητικά έξοδα, οι διοικητικές δαπάνες. Ευχαριστούμε κυρία Εκ. Λοιπόν, τώρα... Δημόσθενες Χάρα, έχεις το λόγο. Πρόεδρε, χτες ο κύριος Ανδροπάου, ο πρόεδρος του Συμβουλίου, είπε ότι δεν είναι δυνατόν να είναι κανείς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Εντάξει, βέβαια, αλλά πηγαίνουν, περνάμε από την Ορβηγία, από την Ελβετία. Κοιτάξτε, ο σύγχρονος πατριωτισμός βασίζεται στην καταστροφή άλλων χωρών. Όχι όμως, διότι υπάρχουν πολλές χώρες που αναγνωρίζουν την ε, δημοκρατία, τα δικαιώματα των άλλων χωρών. Και όταν έφτασε στο δεύτερο σημείο του για τον ευρωσκεπτικισμό που τον προσωμείωσε με τον εθνικισμό και τον πόλεμο, ας ε, μην ξεχνάμε γιατί έγιναν οι πόλεμοι που έγιναν για την ελευθερία, την ελευθερία όλων των χωρών εξαιτίας πατριωτισμού. Η κυριαρχία, η ανεξαρτησία επανακτήθηκαν και βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Ιδιαίτερα σήμερα πρέπει να το θυμόμαστε αυτό. Καλώς κύριε Χάρα. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε και περνάμε στην διάσκεψη Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών και το λόγο έχει η κυρία Αντρέα Κενέφη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ καλωσορίζω την απόφαση του Προέδρου Μπαρακ Ομπάμα να παρακολουθήσει την διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΠΑ ε, αυτό το μήνα στη Λισαβόνα. Υπάρχουν τόσα πολλά σημαντικά θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Η ατζέντα Ένωσης ΙΠΑ ε, είναι πληρέστατη και τα δύο μέρη θα πρέπει να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να προωθήσουν κοινέ θέσει για θέματα όπως οι χρηματοπιστωτικοί κανονισμοί, οι αλλαγές κλιματικές ε, και καταπολέμηση της τρομοκρατίας, οικονομική ανάκαμψη ωστόσο θα πρέπει να είναι το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Η οικονομική μας συνεργασία είναι βασική κινητήριος δύναμη της παγκόσμιας ε, οικονομικής ευημερίας. Μαζί οι οικονομίες μας αναστοιχούν στο ίμιση της παγκόσμιας οικονομίας και γι' αυτό και πρέπει να βρούμε κοινέ στρατηγικές και δράσεις ώστε να εξασφαλίσουμε σταθερή ανάκαμψη από την κρίση συμπεριλαμβανομένη ε, της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών, πακέτα κινήτρων και στρατηγικές ώστε να αντιμετωπίσουμε σωστά την ε, κερδοσκοπία με τις συναρματικές ισοτιμίες. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Κράης. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή μιλάει και για την μετανάστευση, η οποία τον τελευταίο καιρό έχει οδηγήσει σε καταστροφές και με κοινωνικές και οικονομικές συνήπιες. Και εμείς τι κάνουμε, αποφασίζουμε περισσότερο ακόμα μετανάστευση να φέρουμε από το εξωτερικό στην Ευρώπη. Ιδιαίτερη η παράγραφος 110 είναι πολύ κοινική που λέει ότι η βάση για την μετανάστευση είναι ανεξάρτητοι από ό,τι πληροφορίες έχουμε για αυτούς. Τι θα πει ο κοινό άνθρωπος. Είναι μια προπαγάνδα για κάτι το οποίο έχει αποτύχει εντελώς που είναι μαζική μετανάστευση. Όλες οι πληροφορίες για την πολιτική μετανάστευση πρέπει να αναλυθούν σε βάθος. Και ακριβώς αυτό δεν θέλει το λόμπι υπέρ της μετανάστευσης. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό, κύριο Σκίνερ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι κάπως μπερδεύτηκα με το θέμα του ψηφίσματος της Διασκέψεως Κορυφής Ευρωπαϊκής Ενώσεως και είπα, Πιστεύω ότι το ψήφισμα αυτό είναι πολύ μακροσκελές, δεν λύνει τα προβλήματά μας. Πρέπει να διαχωριστεί κατά τρόπον ώστε τα τεχνικά θέματα του Οικονομικού Συμβουλίου να περιληφθούν σε ένα πρόγραμμα τριών σημείων για να μπορούμε να ε, <clears throat> τα απευθύνουμε στους συναδέλφους στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Επίσης όσον αφορά το εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να τονίσουμε πού μπορούμε ε, να ε, προχωρήσουμε και να προωθήσουμε την κατάσταση και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη γεωργία και τέλος δεν πρέπει να περιμένουν να μας καθορίσουν η μερίσια διάταξη, πρέπει να το πράξουμε εμείς. Βεβαίως ξέρω ότι διαπραγματευόμαστε, αλλά γι' αυτό και το πρόγραμμα έχει αδυναμίες και θα πρέπει να προσβλέψουμε στο νέο κογκρέσο και να μιλήσουμε με τους ομολόγους μας κατά τρόπον ώστε να έχουμε μία πιο αίσια έκβαση στο μέλλον του θέματος. Ευχαριστώ. Κύριε Σκίνερ. Κύριε Κλάς, διαδικαστικό, τι έχει θέλετε. <clears throat> Πρόεδρε, έκανα λάθος στην έκθεση, γιατί είχα γραφτεί δήλωση για τη διάσκεψη κορυφής αυτής Ευρωπαϊκή Ένωση, είπα, και ήταν για άλλο θέμα η επεξήγηση που έκανα. Για ποια έκθεση δηλαδή ήταν η δήλωση που κάνατε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. ήμουνα κατά της παραγράφου 14 όσον αφορά την ε, Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης είπα, που λέει ότι πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας όσον αφορά την ε, λύση του Κυπριακού και της ομιλής μεταξύ Τουρκίας, ε, Κύπρου και Ελλάδας. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει παράνομη κατοχή στην Βόρεια Κύπρου από την Τουρκία. Και γιατί ζητάμε από τι πολιτείε να παρέμβουν. Οι ΗΠΑ δεν έχουν καμιά σχέση με αυτό. Αντίθετα, η ανάμειξη των ΗΠΑ στήριξε το όλο θέμα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να μιλάμε για μια ομοσπονδιακή Κύπρο και αυτό πρέπει να είναι προϋπόθεση ε, προηγουμένως να έχουν αποσυρθεί τα στρατεύματα της Τουρκίας από την Κύπρο. Αυτό πρέπει να λέμε και όχι να αναγνωρίζουμε de facto την κατοχή της Βόρειας Κύπρου και να ανοίγουμε την ε, πόρτα για μεγαλύτερες ακόμα καταχρήσεις από πλευράς της Τουρκίας. Ευχαριστούμε κύριε Κλάις. Κοιτάξτε, τώρα μιλάμε για την, ε, τις καταστάσεις για το ονόματα των επιβατών. Έτσι, η κυρία Άντρια Κένεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα. Γιατί κατά την άποψή μου το Ευρωκοινοβούλιο οφείλει να δείξει ότι θεωρεί τα θέματα της ασφάλειας, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του οργανωμένου και διεθνούς εγκλήματος ε, πολύ σοβαρά. Όπως επίσης παίρνει πολύ σοβαρά τις σχέσεις με τους εταίρους όπως είπα, ο Καναδάς και η Αυστραλία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει τώρα να συμφωνήσει για την ε, σύμβαση για τη μεταφορά των ε, ομονομάτων των επιβατών, στοιχείων μάλλον των επιβατών και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την δυνατότητα πολύ συνετά. Εφόσον ε, στις 6 Μαου το Κοινοβούλιο είχε αποφασίσει να αναβάλει την ψηφοφορία λόγω τη αίτηση για συνένεση με τις, για τι συμφωνίε με την ΣΥΠΑ και την Αυστραλία καθώ και την ε, συμφωνία με τον Καναδά η οποία δεν ισχύει πια για το PNR θα πρέπει να φροντίσουμε ότι με τις συμφωνίες αυτές θα βελτιώσουμε την ασφάλεια στον, ε, στην διδατική περιοχή αλλά και πέρα από αυτή. Και τώρα περνάμε στο σημείο της, ε, των συμπράξεων καινοτομία. Το λόγο έχει για ένα λεπτό και ο Σκάσμαρκ. Ευχαριστώ. Ε, είναι ένα πολύ βασικό πρόγραμμα για την Ευρώπη και στο πώς να ε, ε, οργανώθηκε μία διεθνής συνάντηση επί του θέματος αυτού και θα πρέπει να υπάρξουν συντονισμένες προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα περιφερειακό, ευρωπαϊκό, τοπικό για να προχωρήσουμε. Γι' αυτό και υπερψήφισα αυτή την έκθεση διότι πιστεύω ότι η καινοτομία είναι πολύ βασική για το μέλλον μας. Για τον ΟΑΣΕ, κυρία Ανδρίκενον, για ένα λεπτό. Νομίζω ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον οργανισμό είναι πολύ σημαντικός για να επιτευχθούν οι στόχοι. Η Ένωση επιπλέον και ο Ασεαν και είναι διαφορετικές δομές, ε, καθοδηγούνται από τις ίδιες αρχές και αξίες, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατία. Υποστηρίζω τη διάταξη αυτή του κανονισμού όσον αφορά ε, του ψηφίσματος, συγγνώμη, όσον αφορά το Καζακστάν, ώστε να προβούμε σε βήματα για να στηρίξουμε τις βασικές αρχές ε, της ΟΑΣΕ, δηλαδή σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, ελευθερία έκφρασης και όταν θα γίνει εκεί η σύνοδος του ΑΣΕ να γίνει χωρίς εμπόδια. Αυτή Αυτός ο οργανισμός αποτελείται από κράτη που στηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αξίες και θα πρέπει να αποτελεί υπόδειγμα για τις υπόλοιπες χώρες. Ευχαριστώ τώρα για τη δημογραφική πρόκληση η κυρία Νέβε Δαλόμπα. Ε, δεν είναι στην αίθουσα. Η κυρία Ρονσούλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα γιατί θεωρώ ότι προτείνει χρήσιμε και ενδιαφέρουσε προτάσει για να αντιμετωπίσουμε τι μελλοντικέ δημογραφικέ προκλήσει. Οι κοινωνικέ πολιτικέ των κρατών μελών θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στου νέου, που είναι μια πραγματική κινητήριο δύναμη τη ανάπτυξη και τη ε, ε, εξέλιξη. Θα πρέπει να ευνοηθεί η είσοδο των νέων στην αγορά εργασία μέσω μόνιμη κατάρτιση ε, και η οικογένεια θα πρέπει να προστατευτεί με πιο κέρια μέτρα και πιο συγκεκριμένα μέτρα. Γιατί αν ξεχάσουμε την οικογένεια σημαίνει πως εγκαταλείπουμε ένα από τα σημαντικά στοιχεία της κοινωνίας. Ε, υπογραμμίζω λοιπόν τη σημασία των παραγράφων που περιλαμβάνουν μέτρα που είναι υπέρ της ε, οικογένειας Επιπλέον, για να μπορούμε να συγχειριστούμε καλύτερα τις επιπτώσεις της γύρανσης, θα πρέπει να στηρίξουμε την εξυγχρονισμό των κοινωνικών συστημάτων πρόνοιας και των συνταγματικών ε, καθεστώτων. όπω έλεγε ο Σπινέλη, το να φτιαχτεί η Ευρώπη εξαρτάται και από σένα. Και τώρα είναι μια συγκεκριμένη δυνατότητα που έχουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καλινόφσκι. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι δημοκρατικές αλλαγέ Οι δημογραφικές συγγνώμη, αλλαγές στις τελευταίες δεκαετίες στην Ένωση επεστείνουν την προσοχή μας στην ανάγκη μεταρρύθμιση των κοινωνικών και συνταξιδοτικών συστημάτων. Επίσης θα πρέπει να εφεύρουμε βιώσιμες βιώσιμα και αποτελεσματικά συστήματα μετανάστευση. Είδαμε κόσμο που συνταξιδοτείται νωρίτερα, πράγμα το οποίο καταλήγει σε μειωμένε επαγγελματικέ δραστηριότητε για τις ε, ηλικίε μεταξύ 55 και 60 ετών. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε πολύ μεγάλη ενεργία στους νέους. Πρέπει λοιπόν να στηριχθούν οι άνθρωποι από διάφορες ηλικιακέ ομάδες ώστε να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας. Χρειάζεται καλύτερη μεταναστευτική πολιτική και, ε, ε, ε, και πολιτική ένταξη των μεταναστών για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το προβλήματα της γυράσκουσας κοινωνίας. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό ο κύριος Κασμάρεκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε σχετικά με... Θα ήθελα να αναφερθώ στην έκθεση αυτή για τις δημογραφικές προκλήσεις. Πιστεύω ότι η έκθεση είναι καλή και προωθεί σημαντικά θέματα. Ουσιαστικά δεν πρέπει να υπάρχει διάκριση από πλευράς ηλικίας και θα πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη. Είναι ένα βασικό θέμα να υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των γενιών. Δεν πρέπει οι πιο ηλικιωμένοι να την χάνουν κάνουν διακρίσεως επειδή ε, ε, για λόγους ηλικίας και να επικεντρώνουμε την προσοχή μας εις την νεολαία μόνο. Αυτό είναι καλό μεν, αλλά από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να ξεχνούμε και αυτούς οι οποίοι έχουν πολύ συμβάλει στην οικοδόμηση της Ευρώπης. Κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ. Ε, συμφωνώ με την ε, ε, έκθεση αυτή και το θέμα της αλληλεγγύης που είναι πολύ σημαντικό και στην παράγραφο 24 μιλάμε για υποχρεωτική άδεια συνδεξιοδοτήσεως. πιστεύω ότι θα έπρεπε αυτό να είναι προαιρετικό και να υπάρχει μία ηλικία όπου θα αρχίσει κανείς να λαμβάνει τη σύνταξή του. Ε, στην ε, παράγραφο 25 αναφέρεται το θέμα της περιθράψεως ε, εντός της οικογένειας για να δούμε αν κάποιος μπορεί να τύχει περίθαλψη στο σπίτι του ή να υποφεληθεί εν πάση περιπτώσει πλήρως από τα κοινωνικά συστήματα ασφαλίσεως άλλωστε όσον αφορά την επανεκπαίδευση των μακροχρονίων ανέργων θα πρέπει να την προωθήσουμε διότι στην τωρινή κατάσταση της οικονομίας η αλληλεγγύη είναι βασική μεταξύ των γενεών. Η κυρία Μορκουνάιτε τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τη έκθεση του Τόμα Μαν, διότι αντιπροσωπεύει και την αλληλεγγύη και την επαφή ανάμεσα στις γενναίες. Συνήθως μιλάμε για τα δημογραφικά προβλήματα της Ένωσης και το ρόλο της νεότητας. Όμως αυτό το έγγραφο καλύπτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όλων των γενναών, καθώς και τα σχετιζόμενα προβλήματα στον τομέα της απασχόλησης, στον τομέα της υγειονομική περίθαλψης και ούτω καθεξής. αναζητάμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Οι γενναίες Φυσικά θα πρέπει να είναι ευγνώμονες για, να, είναι για την συμβολή τους και η Η γύρανση, θα πει, ή μάλλον οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να λαμβανθούν σοβαρά υπόψη, όμως θα πρέπει να δούμε μέσω των εκπαιδευτικών συστημάτων και να αναπτύξουμε μάλλον περισσότερο τις νέες γενναίες, καθώς και να ενσωματώσουμε τις νέες γενναίες στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χάναν. Κύριε Πρόεδρε, οι ειδικοί περιδημογραφείς μας λένε ότι για να διατηρηθεί ένας πληθυσμός χρειάζεται 2,1 ε, ε, ε, γένες ανά γυναίκα. Στη μόνη χώρα, η μόνη χώρα που λειτουργεί έτσι είναι η Αλβανία ή η Τουρκία, αν την υπολογίσουμε ως ευρωπαϊκή χώρα στην Ένωση. Πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Και η Ρωσία προσπαθεί υπολογίζεται ότι θα χάσουν 100 εκατομμύρια κόσμο τα επόμενα λίγα χρόνια. Η Γερμανία μόνο θα συρρυκνωθεί κατά 20 εκατομμύρια. Αυτά δεν είναι προεκβολέ του τι θα γίνει αν δεν κάνουμε κάτι. Είναι αυτό που θα συμβεί ούτω ή άλλω. Η παρακμή στη γεννητικότητα υπάρχει, η μείωση στη γεννητικότητα υπάρχει. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει μετά από αυτή την ε, προθεσμία. Τι, γιατί έγινε αυτό, τι συνέβη στο παρελθόν. Πολλά γίνονται, πολλά, σε πολλά οφείλεται, υπάρχει αντισύλληψη, υπάρχει ο διαφορετικό ρόλο των γυναικών στην κοινωνία, η μακροζωία, αλλά διερωτώ με μήπω ένα μέρος του προβλήματος είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει επεκταθεί το κράτος και έχει ε, ε, ε, εξορίσει την ιδιωτική σφαίρα ας πούμε, φροντίδα για τα παιδιά, κοινωνική ασφάλιση, ενώ η πρώτη γενεά που, που, που λειτουργήσε με πλήρη κοινωνική περίθαλψη από το λίκνο μέχρι στον ε, τάφο, είναι αυτή η οποία επέφερε αυτή τη μείωση της γεννητικότητας. Ένα σωρό κόσμος πρέπει να δουλεύει για να πληρώσει τα συντάξεις, τις συντάξεις. Θα πρέπει να είναι ένα σύντημα τη πρώτη προτεραιότητα και δεν πρόκειται να ρυθμιστεί μόνο με αυτού του κανονισμού απασχόληση. Περνάμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Καρβάλιο για την απλοποίηση και εφαρμογή των προγραμμάτων πλαίσιο έρευνας. Για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Πέσατς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζω την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή να απλοποιηθούν τα ερευνητικά προγράμματα. Χάρη στην απλοποιημένη μέθοδο θα είναι εύκολο να, ευκολότερο να έχει κανείς χρηματοδότηση αλλά έχει αυξηθεί και η γραφειοκρατία. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα νέο σύστημα το οποίο θα είναι διάφανο όπου θα λαμβάνονται οι υπόψη και θα απλοποιούνται και οι ε, διοικητικές διαδικασίες. Βεβαίως όλα αυτά συνεπιφέρουν ορισμένους κινδύνους αλλά ένας καλύτερος έλεγχος αυτών των δημοσιονομικών μηχανισμών οδηγεί σε μία δυσκινησία του συστήματος και ε, θα πρέπει να ε, έχουμε υπόψη μας αυτό όταν μιλάμε για το 7ο και 8 το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και την προετοιμασία του 8ου προγράμματος πλαισίου. Ευχαριστώ. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι επένδυση και καινοτομία, για να έχουμε καινούριε τεχνολογίες. Για να επενδύσουμε στις ε, νέες τεχνολογίες θα πρέπει να επενδύσουμε και στην έρευνα και αναφέρομαι στα ερευνητικά προγράμματα πλαίσιο τα οποία είναι μοναδικά ανά τον κόσμο και μόνο με αυτή την έρευνα θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Ξέρουμε τώρα ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε επιπλέον θέσεις εργασίας και να βελτιώσουμε το βιωτικό επίπεδο όλων των Ευρωπαίων. Θα πρέπει λοιπόν να ε, ε, διαμορφώσουμε για τις κατάλληλες διοικητικές διεργασίες, δηλαδή καλύτερη πρόσβαση στην έρευνα και γι' αυτό υπερψήφισα αυτή την έκθεση. Τώρα ο κύριος Πυρίλο. Facilitare l'accesso al sistema η διευκόλυνση στην πρόσβαση συστήματος ε, στήριξης που προβλέπεται για το πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας σημαίνει μεγάλη όθηση γιατί δυνατό, στις δυνατότητες ε, ανταγωνιστικότητας ολόκληρου του παραγωγικού συστήματος Ευρώπης. Με τη σημερινή ψηφοφορία είμαι πεπισμένος ότι συμβάλαμε σημαντικά στην επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου, κυρίως για το σύστημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας όλων των κρατών μελών. Συχνά αυτοί, αυτές δεν μπορούν παρά την υψηλή ποιότητα της παραγωγής τους να έχουν πρόσβαση με ευκολία στους απαραίτητους πόρους ώστε να αυξήσουν ακόμη περισσότερο τα παραγωγικά του στάνταρ. Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε όπως το έκανε και η συγκήτρια, πως η ψηφοφορία ήταν ε, σκόπιμη και κέρια γιατί πρόκειται να γίνει η ενδιάμεση αξιολόγηση του 7ου προγράμματος πλαισίου και ευχαριστούμε λοιπόν την εισηγήτρια για τη δουλειά της. Ευχαριστώ, σας ευχαριστούμε κύριε Πύριλο. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Μορκουρέιτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα το έγγραφο για την απλοποίηση της των ερευνητικών προγραμμάτων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και έχασα μέγα τμήμα της συζήτησης στην Ολομέλεια. Το έγγραφο το ίδιο είναι πολύ σημαντικό και η υιοθέτησή του είναι πολύ, πολύ θετικό βήμα. Είναι πολύ σημαντικό όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να μπορούν να συμμετέχουν στο πλαίσιο ε, έρευνας, ε, στα κοινά προγράμματα τα ερευνητικά, γιατί δεν είναι θέμα μεμονωμένων κρατών, πρόκειται για το συμφέρον των κρατών μελών. Όλα τα κρατημέλη έχουν προτιμήσεις Είναι γι' αυτό απαραίτητο να εξασφαλιστεί αμερόληπτη επιλογή και χρηματοδότηση για όλους τους επιστήμονες, όλους τους ερευνητές, γιατί η επιστημονική πρόοδος ε, παράγει προστιθέμενη αξία ε, και οι μη κερδοσκοπικοί επιστημονικοί οργανισμοί θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά επιστημονικά προγράμματα και γι' αυτό ήθελα να το καλωσορίσω και με αυτές τις διευκολύνσεις θα προχωρήσουμε πολύ. Ωραία, περνάμε τώρα στην κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας. Για ένα λεπτό το λόγο έχει η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος είπε ότι θέλει να κοιτάξει την ε, στήριξη της αγοράς όταν είναι αναγκαία. Ναι, αλλά πρέπει να έχουμε κάποια βεβαιότητα για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι δέχονται επιθέσεις από κάθε πλευρά, από την αύξηση των τιμών, από την κερδοσκοπία. Είδα ότι εγκρίθηκε η τροπολογία αυτή που ζητάει τον Επίτροπο να ασχοληθεί αμέσως με το θέμα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στα εισαγόμενα προϊόντα. Τουλάχιστον κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Ακούσαμε επίσης και το υψηλό κόστος της συμμόρφωσης για να έχουμε οι ε, ίδιες συνθήκες. Το ελεγκτικό συνέδριο, μην ξεχνάμε, ότι έχει ετοιμάσει την έκθεσή του και αναφέρεται στη ζάχαρη και, και μία από τι συστάσει που κάνει είναι ότι η διαμόρφωση των τιμών πρέπει να ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι αγώνε ανταγωνισμού τίθενται σωστά σε εφαρμογή στον τομέα αυτό για να έχουν και οι καταναλωτέ σωστέ τιμέ. Αυτό πρέπει να το κάνουμε όχι μόνο στη ζάχαρη, σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα. Ευχαριστούμε κυρία Χάρκιν. Ένα λεπτό τώρα κύριο Σπύρν. Ευχαριστώ. Είμαι υπέρ της πρότασης ψηφίσματος, γιατί εδώ και χρόνια διαπιστώνουμε στην Ευρώπη τη μία κρίση μετά την άλλη, σε βάρος της κτηνοτροφίας, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους κάθε φορά. είτε πρόκειται για την εισαγωγή βόηου κρέατος, αίγιου, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι πλήττουν την κτηνοτροφία. Όπως επίσης και την γαλακτοκομία. Και αυτό είναι η αστάθεια στις τιμές των δημητριακών. Εν ώψη λοιπόν της ΚΑΠ μετά το 2013, καλό θα ήταν να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και να βρούμε μέτρα ώστε για όλον τον γεωργικό τομέα να περιορίσουμε την αστάθεια στις τιμές. Καλό λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει να αντιδράσει γρήγορα για να αντιμετωπιστεί όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτή η κατάσταση κρίσης. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Κέλλη. Παρακαλώ κύριε Κέλλη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι υπέρ της έκθεσης αυτής και χάρηκα που άκουσα τον Επίτροπο σήμερα το πρωί. Πρώτα απ' όλα, η έκθεση του λεκτικού συνεδρίου χτες δείχνει ότι μετά από 1,2 εκατομμύρια αντιστάθμιση και πολλές ε, απώλειες σε θέσεις εργασίας έχουμε 25% μόνο αυτάρκεια. Παρακολούθησε ένα σεμινάριο για την Γεωργία εδώ και εκεί τα ίδια άκουσα. Η αλία, στην αλία τα ψάρια από το Βιετνάμ μας έρχονται. Σε όλους τους τομείς διαπιστώνουμε ότι άλλες χώρες εξάγουν προϊόντα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το κάνουν με πολύ πιο συμφέρουσες οικονομικά συνθήκες από ό,τι μπορούμε εμείς να παράγουμε και να εξάγουμε τα δικά μας προϊόντα. Πρέπει να υπάρχουν ίδιες προδιαγραφές να ισχύουν τα ίδια για προϊόντα που έρχονται από τρίτες χώρες στην Ευρώπη, όπως ισχύουν και για τα προϊόντα που έχουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, τίποτα άλλο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τις επεξηγήσεις ψήφου. Τα πρακτικά θα υποβληθούν προς έγκριση στο σώμα στην αρχή της επόμενης ε, συνόδου.